την άλλη επόμενη Συνόδου Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, θα προωθήσω τα εγκεκριθέντα σήμερα ψηφίσματα στους αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στα ψηφίσματα. Διακόπτεται η συνεδρία.